Buon Καθίστε παρακαλώ για να ξεκινήσουμε τις εργασίες της Επιτροπής μας. Καταρχάς, να υιοθετήσουμε το σχέδιο ημερησίας διάταξης με μία τροποποίηση να αναβάλουμε την ε, παρουσίαση της μελέτης για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Σύλλου. Αν δεν υπάρχουν ε, αντιρρήσεις, εγκρίνεται η μερίσια διάταξη. Δεύτερον, ανακοινώσεις του Προέδρου. Δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Ωστόσο, θα ήθελα απλώς να σας ενημερώσω ότι η διάσκεψη των Προέδρων των Πολιτικών Ομάδων ανέθεσε στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών να οργανώσει μια έκτακτη συνεδρίαση με την Αντιπρόεδρο, την κυρία Ρέντινγκ, και τους Επιτρόπους ε, Μάλστρομ και Άντερ για να συζητήσουν τη συνέχεια που θα πρέπει να δοθεί στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου που υιοθετήθηκε στην Ολομέλεια προσφάτως για το θέμα των ε, Ρωμά το οποίο συζητήθηκε και στην ε, ε, Σύνοδο Ολομελία του Στρασβούργου σε μια συγκεκριμένη συνεδρίαση συντονιστών που οργανώθηκε ακριβώ για αυτό το σκοπό. Σημειώστε λοιπόν ότι αυτή η συνεδρίαση θα γίνει την Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου στις 4. Προτείνω τώρα να εγκρίνουμε την πρόταση των συντονιστών για τους ε, εισηγητές για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Έρευνας, ο κύριος Μέλο, για τις ε, την εποχιακή εργασία ο κύριος Μωράες, η Ακολίνο για τις πολυεθνικές, Ευρωπαϊκή Στρατηγική κατά της τρομοκρατίας, Σοφία Τουέλ. Και να σας υπενθυμίσω επίσης ότι αύριο το απόγευμα και μεθαύριο το πρωί θα γίνει στα πλαίσια της έκθεσης Αντζελίλη μία ακρόαση με θέμα την καταπολέμηση της ε, σεξουαλικής βίας κατά των παιδιών. Ο κύριος Κλάης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μόλις μας παραπέμψατε στη συνεδρίαση των συντονιστών της Επιτροπής μας που έγινε στο Στρασβούργο την περασμένη Τρίτη παρουσία της Επιτρόπου Μάρσρομα και της Επιτρόπου Ρέντινγκ. Ε, ε να προετοιμάσουμε και επόμενες συνεδριάσεις. Αλλά γιατί, θέλω να ρωτήσω τώρα, πριν τη συνεδρίαση της Τετάρτης πρέπει να γίνει και άλλη συνεδρίαση ε, στο Στρασβούργο των συντονιστών. Κανονικά ούτε αρμοδιότητα είναι ούτε στόχος ε, τέτοια συνεδρίαση των συντονιστών. Ο κανονισμός του Κοινοβουλίου ορίζει ότι συνέρχονται οι συντονιστές για να ρυθμίσουν θέματα ε, διαδικαστικά και να μοιράζουν εκθέσεις στι πολιτικές ομάδες. Τι σχέση έχει αυτό τώρα με αυτά τα θέματα τα δύο, ούτε με το ένα ούτε με το άλλο. Ήταν κατεξοχήν πολιτικού χαρακτήρα και δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο δεν εκλήθησαν όλοι στη συνεδρίαση αυτή, δηλαδή και μία εγγεγραμμένη, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Μας απαγόρευσαν την είσοδο στη συνεδρίαση των συντονιστών. Απαράδεκτα πράγματα για μένα. Το θέμα των Ρωμά ήταν ένα ζήτημα το οποίο συζητήθηκε επί μακρόν, ήταν και πολύ περίπλοκο και προέκυψε από μια συγκεκριμένη επιλογή που έκανε η πρόεδροι των πολιτικών ομάδων, δηλαδή ζήτησαν από την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών να συζητήσει το θέμα αυτό και αυτό θα κάνουμε την επόμενη Τετάρτη στις 4 και θα σταθούμε και στους λόγους για τους οποίους δεν συμπεριλήφθηκε η ομάδα σας. Θα το συζητήσουμε στην συνεδρίαση με τους συντονιστές που θα γίνει αύριο το πρωί. Στο σημείο 3 τώρα της ημερήσιας διάταξης και σημείο έχουμε δύο σχέδια συμφωνίας με τη Γεωργία που αφορούν την επανεισδοχή προσώτων που διαμένουν χωρίς άδεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων. Να ζητήσω λοιπόν από την κυρία Γκρίσμπεκ, η οποία είναι η εισηγήτρια για τα θέματα αυτά, αρχικό στο λόγο και στη συνέχεια θα παρέμβουν όσοι από τους αδέλφους θέλουν να ε, ε, παρέμβουν και στη συνέχεια θα ακούσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η εισηγήτρια παρακαλώ. Mes chers collègues, Αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Αν συμφωνείτε, θα ήθελα να κάνω κοινή την παρουσίαση των δύο σημείων που αφορούν την επανεισδοχή ανθρώπων που είναι, παραμένουν εδώ παράνομα και την πρόταση συμφωνίας που στόχο έχει τη διευκόλυνση της ε, χώρισης θεωρήσεων. Αυτά τα δύο κείμενα, αυτά τα δύο θέματα που έχουν υποβληθεί προς έγκριση για μας και εσείς συμβουλεύω να τα εγκρίνετε, ε, πηγαίνουν χέρι-χέρι. Επιτεύχθηκε συμφωνία για την προηγούμενη εβδομάδα για το Πακιστάν, για την πανεισδοχή ανθρώπων πολιτών του Πακιστάν. Ε, αυτό μου δημιουργούσε πρόβλημα, ενώ εδώ μιλάμε για εταιρική σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γεωργίας και τα πράγματα είναι πολύ πιο σαφή. Ε, δύο λόγια να σας πω για, σύντομα για να σας παρουσιάσω το θέμα. Μετά από την σύραξη τον Αύγουστο 2008 στη Γεωργία υπήρξε ένα έκτακτο συμβούλιο κορυφή που συνεδρίασε το Σεπτέμβριο του 2008 και αποφάσισε την ε, σχέση, να, να τονώσει τη σχέση μεταξύ Ένωση και Γεωργία, κυρίω μέσω τη διαδικασία απλοποίηση τη διαδικασία εκχώρηση θεωρήσεων. Υπήρξε αρχικά μια συμφωνία με στόχο τη διευκόλυνση της εκχώρησης ε, θεωρήσεων, αλλά ε, με την προϋπόθεση ότι θα υπέρχει και συμφωνία Σε Τον Νοέμβριο του 2008 ε, το Συμβούλιο έδωσε την εξοδότηση στην Κομισιόν να διαπραγματευτεί τη συμφωνία αυτή και έτσι είχαμε ένα σχέδιο κειμένου που να πλαισιωθούν οι αρχές που θα διέπουν αυτές τις διαδικασίες και είχε δημιουργηθεί και ένα σχετικό πλαίσιο συνεργασίας ε, και διαπραγματεύσεων με τις γεωργινές αρχές. Το 2009 υπογράφηκε ένα αρχικό κείμενο από τους διαπραγματευτές των δύο πλευρών. Είναι σαφές ότι το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία επιθυμούν να συμμετέχουν στη συμφωνία και άρα επιβαλόταν μια προθεσμία τριών μηνών πριν από τη συνυπογραφή της συμφωνίας. Ε, επιχρεώσεις σε θέματα επανεισδοχής, αυτά όλα βασίζονται σε μια απόλυτη αμοιβαιότητα και οι διατάξεις ισχύουν τόσο για τους ε, υπηκόους ε, της Ένωσης όσο και για τους υπηκόους τρίτων χωρών. Η επανεισδοχή των, ε, των υπηκών της Ένωσης συμπεριλαμβάνει και πρώην υπηκόους που είχαν εγκαταλείψει την εθνικότητά τους ή που είχαν γίνει δεκτοί χωρίς να πάρουν την εθνικότητα κάποιου άλλου κράτους. Και Εκεί καλύπτονται και τα μέλη της οικογένειας, ε, όποια και αν είναι η εθνικότητά τους. Η συμφωνία ορίζει τις διαδικασίες επανεισδοχής, δηλαδή το ενέτηση επανεισδοχής, ε, τα ε, έγγραφα που χρειάζονται, οι προθεσμίες που ισχύουν, η μεταφορά, διαδικασίες διέλευσης και όλα αυτά που σχετίζονται με τις διοικητικές διαδικασίες γύρω από αυτή την συμφωνία. Καθώς και θεσπίζει και εγκαθιδρύει όπως σε όλες τις συμφωνίες επανεισδοχής μια επιτροπή Μικτή Επιτροπή επανεισδοχής που θα αποφασίσει για τον εσωτερικό της κανονισμό. Να σας θυμίσω ότι και υπογραμμίστηκε την περασμένη εβδομάδα στην Ολομέλεια στο Στρασβούργο ότι για την ώρα για τις συμφωνίες επανεισδοχής δεν έχουμε καμία αξιολόγηση όσον αφορά την εφαρμογή τους και ότι προφανώς στο πλαίσιο αυτών των δύο συμφωνιών επιθυμούμε Επιθυμούμε να έχουμε αξιολογήσεις όσον αφορά την εφαρμογή των συμφωνιών επανεισδοχής, τουλάχιστον για αυτές που έχουν ήδη αρχίσει να ισχύουν. Υπογραμμίζουμε επίσης και στα δύο κείμενα την βούληση να καταλήξουμε σε πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και βεβαίως σύμφωνα με τα διεθνή ισχύοντα μέσα που αφορούν αυτόν τον νομικό τομέα. Να υπογραμμίσουμε επίσης σε σχέση με τις σημαντικές συζητήσεις που είχαμε την περασμένη εβδομάδα για την ε, Συμφωνία Επανεισδοχής που την περασμένη εβδομάδα, όπως σας είπα, ε, εντάξει, τα έχουμε ήδη πει, αλλά ας το ξαναπώ, ε, ήταν η πρώτη συμφωνία επανεισδοχής στο πλαίσιο της συνθήκης της Λισαβόνας. Δεσμεύουμε λοιπόν την ευθύνη μας ακόμη περισσότερο από νομικής και από πολιτικής άποψης για όλες τις υπόλοιπες συμφωνίες, διότι είμαστε συν ε, νομοθέτες και θυμίζω για να διαφοροποιηθούμε από τη συμφωνία της περασμένης εβδομάδας ότι αυτές οι δύο συμφωνίες έγιναν με μια χώρα που έχει υπογράψει τη Σύμβαση της Γενέβης και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Πράγμα που μας δίνει έναν κάποιο βαθμό εγγύησης πολύ ανώτερο από ό,τι η προηγούμενη υπόθεση. Δύο λόγια για τη δεύτερη συμφωνία που αφορά την διευκόλυνση χορήγησης θεωρήσεων. Για όλους τους ετούντες αυτή η συμφωνία ισχύει. Θα πρέπει η απόφαση για την χορήγηση ή όχι της θεώρησης να λαμβάνεται μέσα σε 10 μέρες, δηλαδή σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα και θα επεκτείνεται μέχρι τις 30 μέρες όταν χρειάζεται κάποια παραπάνω πληροφορία. Σε επίγουσες ε, περιπτώσεις μπορεί να περιοριστεί στις δύο εργάσιμες μέρες. 35 ευρώ θα καταβάλουν οι γεωργιανοί υπήκοοι για να πάρουν ε, θεωρήσεις. Ε, εν πάση περιπτώσει τώρα δεν χρειάζεται να σας πω όλες αυτές τις λεπτομέρειες. Ε, υπάρχουν και διάφορα άλλα διοικητικά στοιχεία τα οποία εδώ στη δεύτερη συμφωνία περιλαμβάνονται και ορίζονται σαφώς. Αυτό φυσικά σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα στον δρόμο για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Για να ολοκληρώσω και να, περάσω, να δώσω το λόγο στην Κομισιόν και στους συναδέλφους να πω ότι αυτή η συμφωνία εντάσσεται σε ένα γενικότερο συνεργασία με του γείτονέ μα προ Ανατολέ Λάς και προ Νότο, με όλε τι χώρε του Νότιου Κάφκασου ε, και πέρα από τη βούληση εμβάθυνση των σχέσεων με αυτέ τι χώρε που βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα τη Ένωση, ο στόχο είναι να προωθηθεί επίση η ασφάλεια ε, μια μορφή σταθερότητας και ανάπτυξης των σχέσεων μεταξύ της Ένωσης και της Γεωργίας. Και άρα όλα αυτά να μπουν σε ένα σαφές ε, νομικό πλαίσιο το οποίο διέπεται από πλήρη αμοιβαιότητα. Αυτά λοιπόν σε σχέση με αυτές τις δύο συμφωνίες κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε την κυρία Γκρίσμπεργκ. Έχει ζητήσει το λόγο η κυρία Φαζόν. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Najprej bi se rada zahvalila Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και για τα δύο έγγραφα και να της εκφράσω την υποστήριξή μου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ακριβώς να ανοίξουν οι θύρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις τρίτες χώρες προκειμένου για τους πολίτες της Γεωργίας βεβαίως ε, εφόσον πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται. Κατά τη διάρκεια του περσινού έτους πράξαμε το ίδιο για τη Σερβία και το Μαυροβούνιο ενώ φέτος για την Αλβανία και τη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το βήμα κατά την άποψή μου για να καταργηθεί κάποια στιγμή η υποχρέωση θεώρησης διαβατηρίου. Έτσι, ώστε οι πολίτες των χωρών αυτών να μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα και ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα εδώ εγώ για τους φοιτητέ που πλήττονται πάρα πολύ περισσότερο από τους άλλους 60 ευρώ κοστίζει η βίζα αντί για 35 και είναι μεγάλη επιβάρυνση αυτή για τους νέους, τους φοιτητέ και τους δημοσιογράφους θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να έρχονται στην Ευρώπη Έτσι θα μπορέσουμε εμεί να έχουμε και πιο στενές σχέσεις και καλύτερη συνεργασία με τη Γεωργία και πολιτιστική μεταξύ άλλων. Κάτι άλλο που θέλω να σας πω αυτή τη στιγμή είναι πάλι σχετικό με τη διευκόλυνση ε, χορήγησης ε, θεώρηση διαβατήριων είναι ο τρόπος με τον οποίο θα εφαρμοστούν όλα αυτά. Ε, οι προηγούμενε χρονίε έδειξαν ότι στα Βαλκάνια δεν είναι αυτόματη η διευκόλυνση, ούτε πραγματικότητα η διευκόλυνση στην πράξη. Μπορεί θεωρητικά να ισχύει, αλλά θα πρέπει να φροντίσουμε να εφαρμοστεί πλήρως και με τον τρόπο που έχει σχεδιαστεί αυτή η διευκόλυνση. Να γίνονται βεβαίω πάντα σεβαστά τα κριτήρια. Δεν αντιλέγω. Και κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Θα πρέπει να γίνει και απαραίτητη ενημερωτική εκστρατεία για να γνωρίζουν οι πολίτες τι σημαίνει αυτό. Για να μην υπάρξουν παρεξηγήσεις. Δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση για ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών αυτών των χωρών διότι παραμένουν ακόμα κάποιες προϋποθέσεις, κάποιοι περιορισμοί που θα πρέπει να γίνονται σεβαστοί. Δεν είναι πλήρης ε, απελευθέρωση της κυκλοφορίας των προσώπων αυτό. Το συντομότερο λοιπόν, αυτή τη στιγμή είναι έτοιμα και τα ίδια τα κράτη, ε, θα πρέπει να είμαστε και εμείς σε θέση να καταργήσουμε τα διάφορα εμπόδια, είτε αυτό είναι τεχνικής φύσεως, είτε ό,τι έχει να κάνει, όπως σας είπα, με την εφαρμογή, με την υλοποίηση και την πολιτική πτυχή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στο βαθμό του δυνατού θα πρέπει να φροντίζει να έρχεται πιο κοντά στους γείτονές της και οι γειτονικέ χώρες να έχουν την ευκαιρία να συμμερίζονται τις αρχές και τις αξίες μας. Και ιδιαίτερα ναι, ευχαριστώ και πάλι την εισηγήτρια και είμαι στο πλευρό σας. Ευχαριστώ. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. E, Κύριε Πρόεδρε, δεδομένου ότι η κυρία Γκρισμπέκ σε αυτή την εξαίρετη εκθεσή καθώς και οι προηγούμενοι ομιλήτρια εξήγησαν όλα τα επιχειρήματα υπέρ της έκθεσης, θα ήθελα να πω ότι στις 15 Σεπτεμβρίου το συζητήθηκε το θέμα στην Επιτροπή ΑΦΕΤ ε, οι δύο σχετικές γνωμοδοτήσεις υιοθετήθηκαν ε, χωρίς καμία αντίρρηση. Υποστηρίζουμε όλα τα επιχειρήματα που παρουσίασαν οι δύο συνάδελφοι και την σύναψη ως εκ τούτου των δύο αυτών συμφωνιών ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Γεωργία. Να συμπληρώσω ένα επιπλέον επιχείρημα, να σας πω ότι είχα δύο φορές την ευκαιρία να βρεθώ στην Γεωργία μέσω της αντιπροσωπείας της Επιτροπής ΑΦΕΤ και επίση ηγήθηκα τη αντιπροσωπεία τη υποεπιτροπή ΣΕΝΤΕ και γι' αυτό ε, μπορώ να σα πω ότι είχαμε την εντύπωση ότι υπάρχει μεγάλη εξέλιξη στη Γεωργία όσον αφορά το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αυτό ανεξάρτητα από την πολιτική μα προέλευση, από την εθνική μα προέλευση. Να πω ότι εντυπωσιαστήκαμε από την εξέλιξη και την ανάπτυξη του δημοκρατικού συστήματο. Η πρώτη που μου επίσκεψη εκεί αφορούσε την ε, επίβλεψη των εκλογών και διαπιστώσαμε πως η Γεωργία είχε θέσει σε εφαρμογή όλες τις αρχές του κράτους δικαίου με την ε, παρακολούθηση πολλών διεθνών παρατηρητών. Διαπιστώσαμε ότι τηρήθηκαν όλοι οι κανόνες και αυτό είναι πάρα, σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό γιατί ξέρουμε ότι στο παρελθόν είχαν εκφραστεί πολλές επιφυλάξεις. Ε, ε είναι επίσης η προσπάθεια του Προέδρου και της κυβέρνησης όσον αφορά την καταπολέμηση της διαφθοράς στη χώρα αυτή ανεξάρτητα από κάποια εξωτερικά προβλήματα που υπάρχουν υπάρχουν και δεν χρειάζεται να τα συζητήσουμε αυτό τώρα εδώ, θα μπορούσαμε να πούμε πως η χώρα αυτή εξελίσσεται προς τη σωστή κατεύθυνση, αναπτύσσεται ε, σωστά και η Ευρωπαϊκή Ένωση με την υπογραφή αυτών των συμφωνιών θα πρέπει να υποστηρίξει πλήρως τις προσπάθειες της Γεωργίας. Υποστηρίζω λοιπόν τις εκθέσεις αυτής ως συντάκτης των δύο γνωμοδοτήσεων. Σας ευχαριστώ. Ωραία το λόγο έχει τώρα η Προεδρία του Συμβουλίου, η κυρία Ισαμπέλ Ράις. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την εισήγητρια για την παρουσίαση της έκθεσης αυτής που συνάδει πλήρω με την πρόταση Ευρωπαϊκής, ε, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου συγγνώμη, και την θέση του για τις δύο συμφωνίες. Είναι πολύ ε, ικανοποιητικά αυτά και το Συμβούλιο επιθυμεί σύντομα να τεθούν σε ισχύ τα κείμενα αυτά. Ελπίζουμε η διαδικασία να επιταχυνθεί γιατί συμφωνούμε και εμείς ότι χρειάζεται πιο στενή συνεργασία και σχέσεις ε, ενισχυμένες Γεωργίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό θα βοηθήσει και τις διαπροσωπικές σχέσεις ε, επαφές αλλά και την καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης με τη Συμφωνία Επανεισδοχής. Θα δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να παρουσιάσει το περιεχόμενο της συμφωνίας. Θα ήθελα μόνο να σας ε, καθησυχάσω γιατί υπήρξε μια αντίδραση. Δεν είναι απελαγμένοι όλοι οι φοιτητέ από, από την υποχρέωση θεώρησης, αλλά όλα τα παιδιά κάτω των 12 ετών και εκείνοι που συμμετέχουν σε σχολικές εκδρομές. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ο λόγος τώρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κυρία Δάφνη Γόγου έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και την συγκήτρια. Είναι εξαιρετική η έκθεσή της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ικανοποιημένη ε, για την έκθεση και από την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις δύο αυτές συμφωνίες που θα θυμάστε όλοι ότι ε, ακολούθησαν την ταραγμένη περίοδο του 2008 θέλησε η έκτακτη σύνοδος κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Γεωργία να στείλει ένα μήνυμα έντονο. Γι' αυτό και ακολούθησε με αυτή τη ταχύτητα η διαπραγμάτευση και το αποτέλεσμα και των δύο συμφωνιών αντικατοπτρίζει την πολιτική βούληση να προχωρήσουμε γρήγορα έτσι ώστε να ε, τεθούν σε ισχύ οι δύο συμφωνίες. Δεν χρειάζεται να υπενθυμίσω την πολιτική κατάσταση είχαν την ε, καλοσύνη οι αξιότιμοι βουλευτές να το θυμίσουν για τη θεώρηση διαβατηρίων επιτρέψτε μου ε, να πω κάτι σε σχέση με τόσα είπε η κυρία Φαγιών κυρίως οι συμφωνίες διευκόλυνση δεν λαμβάνουν υπόψη μόνο τη θετική εμπειρία που έχουμε αποκομίσει με τις συμφωνίες με άλλες χώρες τη Ρωσία, την Ουκρανία, τη Μολδαβία αλλά και τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων αλλά ε, ε, είδαμε ότι στη συνέχεια εγκρίθηκε και ο κώδικας ε, θεωρήσεων και σε αυτές τις συμφωνίες διευκόλυνσης θεώρησης θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας τα νέα δεδομένα ακριβώς τον κώδικα αυτό και το άρθρο 48 που προβλέπει ενίσχυση της συνεργασίας Σέγγεν σε τοπικό πάντα επίπεδο για να υπάρξει ακόμα μεγαλύτερη εναρμόνιση ε, ως προς τον τρόπο με τον οποίο χορηγούνται οι θεωρείς διαβατηρίων. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται ακριβώς για να διευκολύνει ακόμα περισσότερο τη διαδικασία αυτή να εκπονήσει όπως έκανε για τα Δυτικά Βαλκάνια, κατευθυντήριες γραμμές για το πώς θα εφαρμόζονται ακριβώς αυτές οι συμφωνίες. Τα τελευταία έτη έχουμε καλή εμπειρία από καλές πρακτικές και βάσει αυτών θα ξεκινήσει μια διαδικασία ενημέρωσης, μια ενημερωτική εκστρατεία για να καταλαβαίνουν ακόμα καλύτερα οι γεωργιανοί πολίτες ε, τα νέα δεδομένα και τι ισχύει με τη συμφωνία αυτή. Τώρα, για τη διευκόλυνση των θεωρήσεων να ακολουθούμε την ίδια προσέγγιση όπως και στο παρελθόν. Δηλαδή, διαπραγματευόμαστε και συνάπτουμε τέτοιες συμφωνίες παράλληλα με συμφωνίες ε, επανεισδοχής. Για την περίπτωση όμως της Γεωργίας διαφοροποιήσαμε λίγο ε, τη διαδικασία, όχι την προσέγγιση. Δηλαδή, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία ε, έχουν τη δυνατότητα opting in και για να γίνει αυτό, ε, προτάξαμε λίγο την ημερομηνία υπογραφής της Συμφωνίας Θεώρησης. Πάντως, και οι δύο συμφωνίες θα τεθούν σε ισχύ ταυτόχρονα. Διαβεβαιώνω στην εισηγήτρια ότι μέχρι το τέλη του έτους θα καταθέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, μία πλήρη αξιολόγηση του τρόπου εφαρμογής ε, των συμφωνιών επανεισδοχής που έχουμε υπογράψει μέχρι στιγμής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο Μπρόνς έχει λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όσον αφορά τη Συμφωνία Επανεισδοχής, γιατί θα πρέπει ένα κράτος, η Γεωργία στη δεδομένη περίπτωση, να ε, δεχτεί την επιστροφή τους. Ε, καταλαβαίνω ότι μπορεί να υπάρχει πρόβλημα με τους υπηκόους τρίτων χωρών που ταξιδεύουν παρανόμως στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τη Γεωργία, αλλά νομίζω ότι ε, το λογικό θα ήταν να τους στείλουμε στην τρίτη χώρα και όχι στη Γεωργία από την οποία μας ήρθαν. Ως προς τη διευκόλυνση των θεωρήσεων τώρα. Η διαδικασία αυτή δεν έχει να κάνει με την ε, μετανάστευση και την μόνιμη άδεια παραμονή. Αυτή τη στιγμή κάποιο έχει εισέλθει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχουν κάποιε δικλείδε ασφαλεία, να έχει θέση ασφαλεία ή αλλιώ ε, θα πρέπει να επιστρέψει και δεν θα μπορεί να γίνει μετανάστης επισήμως δυστυχώς είναι ευάλωτη σε εκμετάλλευση οποιασδήποτε μορφής εάν δεν υπάρχει άδεια παραμονής και αυτές οι διευκολύνσεις των θεωρήσεων φοβάμαι ότι δημιουργούν ε, μία, ε, κάτι αντίστοιχο με σχεδόν κράτη-μέλη. Η συγκήτρια τώρα. Euh, euh, Σα ευχαριστώ. Εγώ θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω του συναδέλφου για την ενθάρρυνσή τους και για την έγκρισή τους για τις δύο αυτές εκθέσεις. Να ευχαριστήσω το Συμβούλιο και την Επιτροπή για τις διευκρινήσεις και που έκαναν, καθώς και για το ότι επιβεβαίωσαν την αξιολόγηση, διότι πιστεύω πως η αξιολόγηση είναι πάρα πολύ σημαντική για να μπορέσουμε να τοποθετηθούμε εντός μιας διαδικασίας που θα επιδιώξει τους στόχους που θέλουμε. Και να ευχαριστήσω και τον συνάδελφο Μπρόνς για τις παρατηρήσεις του. Πιστεύω πως είμαστε βασικά, ε, βρισκόμαστε μάλλον αναμονή μιας αξιολόγησης ώστε να μπορέσουμε όχι μόνο για αυτές τις δύο συμφωνίες, αλλά για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε γενικότερα ε, σε σχέση με τις δικές μας γενικές αρχές. Δεν πιστεύω πως ε, υπήρξαν άλλες ερωτήσεις για τους φοιτητές. Ε, οι διατάξεις νομίζω αναφέρθηκαν και πάλι προχωρώντας ε, και μέσω της αμοιβαιότητας αλλά ταυτόχρονα και λόγω του γεγονότος ότι οι δύο συμφωνίες αυτές είναι συνδυασμένες, δηλαδή θεωρήσεις και επανεισδοχή, πιστεύω πως έτσι θα έχουμε ένα ε, υπόδειγμα λειτουργικότητας και καλύτερα είναι να ξεκινήσουμε με αυτό παρά από το Πακιστάν. Ίσως ε, σας κουράζω με την επανάληψη αυτή, αλλά συμβολικά θα ήταν πολύ πιο δυνατή κίνηση όσον αφορά την ε, εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και φυσικά παραμένω στη διάθεση των συναδέλφων να έχουν άλλες παρατηρήσεις. Ευχαριστώ. Καλώς, ευχαριστούμε την εισηγήτρια. Εδώ θα πρέπει να σας κάνω κάποιες ε, ανακοινώσεις σχετικώ με την έκθεση. Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών για τα δύο θέματα που συζητήσαμε. 6 Οκτωβρίου, 12 το μεσημέρι. Και επίσης να τονίσω ότι βάσει της διαδικασίας επιτρέπονται τροπολογίες μόνο για το νομοθετικό ψήφισμα για πτυχές οι οποίες σχετίζονται με τη διαδικασία. Η ψηφοφορία στην Επιτροπή θα γίνει στις 25 και 26 Οκτωβρίου ε, για να συζητηθεί από εκεί και πέρα το θέμα στην πρώτη ολομέλεια του Νοεμβρίου. Έχει ζητήσει το λόγο ο κύριος Κέλλερ. Η κυρία Κέλλερ. Κυρία Κέλλερ, παρακαλώ. Συγγνώμη. Περδεύτηκα. Συγγνώμη που καθυστέρησα. Άλλαξα λίγο το πρόγραμμά μου και καθυστέρησα. Έχω κάποιες ερωτήσεις για την Συμφωνία Επανεισδοχής με τη Γεωργία και με... για τη Συμφωνία για τις θεωρήσεις. Για την επανεισδοχή. γνωρίζει η Επιτροπή ή το Συμβούλιο πόσα άτομα αφορά η συμφωνία αυτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αν γνωρίζουμε για ποιους λόγους ήρθαν. Αν για παράδειγμα ήρθαν ε, κάνοντας αίτηση ασύλου ή για κάποιον άλλο λόγο. Επίσης θα ήθελα να γνωρίζω αν θα σταλούν ε, άτομα στην Απχασία βάσει της συμφωνίας αυτής. Γιατί γνωρίζετε ότι στην περιοχή Ισχύει ακόμα η θανατική ποινή. Επομένως είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Και η Amnesty International και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρόληψη των βασανισμών γνωρίζουν ότι ε, ε, οι βασανισμοί στις φυλακές ε, είναι κάτι ιδιαίτερα διαδεδομένο. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα βίας κατά των γυναικών στη Γεωργία τα οποία περνούν και ατιμόρυτα. Επομένως δεν επιστρέφουν αυτοί οι άνθρωποι σε ιδανικές συνθήκες. Ε, δεν ξέρω αν ε, πρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μπορεί να μας πει κάτι από αυτού. Πρέπει να τη βρω τώρα την ερώτηση που έχω να κάνω για τις θεωρήσεις και να επανέλθω αργότερα. Ζητώ συγγνώμη. Αυτά τα οποία μόλις μας είπατε Μπορείτε κυρία Κέλλερ να τα αποστείλετε με μια επιστολή στη γραμματεία, να ε, παρουσιάσετε την άποψή σας και να λάβετε φυσικά και τις απαντήσεις. Έχουμε ολοκληρώσει τώρα με το θέμα αυτό και να περάσουμε στο επόμενο σημείο, στο σημείο 5. Ελάχιστε απαιτήσει για τι διαδικασίε με τι οποίε τα κράτη-μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώ του πρόσφυγα. Ζητώ τώρα να δώσουμε το λόγο στην κυρία Γκυγιόμ, η οποία θα μας παρουσιάσει το έγγραφο εργασίας της, που σχετίζεται με ένα από τα πιο περίπλοκα θέματα του πακέτου για το άσυλο. Η εισηγήτρια έχει κάνει αρκετέ ε, συναντήσεις με τους κοιόδης εισηγητές και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το θέμα αυτό ε, έχει συζητηθεί επί μακρόν και Φαντάζομαι ότι η συγχύτρια τώρα, στη διάρκεια της παρέμβασής της, θα μπορέσει να μας καθορίσει και κάποιο χρονοδιάγραμμα για το πώς μπορεί να προχωρήσει αυτό το θέμα και ε, θα θέλαμε από το Συμβούλιο που νομίζω ότι δεν έχει κάποιον εκπρόσωπο εδώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας πούν την άποψή της. Κύριε Γιγιόμ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το έγγραφο εργασίας που σας υπέβαλα έχει στόχο ε, να κοιτάξουμε τις ε, σημαντικότερες αλλαγές ε, ε, στην οδηγία του 2005, το έγγραφο εργασίας είναι μακροσκελές αλλά όχι εξαντλητικό. Στόχος είναι να υπάρξει μια πολιτική αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο γίνεται η αναδιατύπωση της οδηγίας θα δούμε και τις τροπολογίες. Πριν μπω στις κατευθυντήριες γραμμές του γράφου, να σας δώσω λίγο το πλαίσιο. Παρά τα μέτρα εναρμόνισης που εγκρίθηκαν τα τελευταία 10 χρόνια για το άσυλο, υπάρχουν μεγάλες ε, διαφορές και παραμένουν από κράτος σε κράτος ως προς την υποδοχή, την ποιότητα ε, της διαδικασίας και τις αποφάσεις. Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Να σας δώσω δύο παραδείγματα. Στα κράτη-μέλη το 2009 η θετική έκβαση 65% μέχρι λιγότερο από 1% σε πρώτο βαθμό. Και εδώ μιλώ για ε, μία χώρα ε, προέλευσης. Τώρα για τη διαδικασία. Την προθεσμία που έχει κανείς για να υποβάλει προσφυγή σε ορισμένες χώρες είναι 30 ημέρες ενώ σε άλλες δύο μόλις ημέρες. Πρόσφατα δημοσιεύθηκαν μελέτες όπως η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται ε, αυτά στα κράτη-μέλη, το δίκτυο Οδύσσεας, η πατιαρμοστία του ΟΗΕ και άλλοι ενδιαφερόμενοι δείχνουν ε, ότι υπάρχουν πραγματικά πολύ μεγάλες διαφορές από χώρα σε χώρα και έχουν να κάνουν με τις χώρες ασφαλούς προέλευσης, ε, τις παλιστρίτες χώρες ε, και τα λοιπά. Αυτές οι διαφορές δεν είναι πολύ συμβατές με ένα κοινό ε, καθεστώς ασύλου που στόχο έχει να είναι αντίστοιχη η προστασία των προσώπων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και έρχεται σε αντίθεση με μία από τις θεμελιώδεις αρχές του Δουβλίνου ότι είναι αντίστοιχα τα συστήματα ασύλου και συγκρίσιμα στα κράτη-μέλη. Μόνο λοιπόν αν υπάρχει εναρμόνιση των ε, δικονομικών εγγύσεων θα ε, υπάρξει πρόοδος. Πρέπει να καταρτιστεί μια λίστα, ένας κατάλογος των χείριστων πρακτικών για να έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είπα, εναρμόνιση των εγγύσεων και των διαδικασιών, των ε, δικονομικών. Το προηγούμενο κείμενο που ήταν μινιμαλιστικό δεν επέτρεψε επαρκέ επίπεδο και ικανοποιητικό εναρμόνιση. και ήταν ει βάρο και της ποιότητα και της αποτελεσματικότητα, της λήψη αποφάσεων, αλλά δεν προστατεύει εκείνου που υφίστανται διώξει. Γενικά θεωρώ ότι η πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή βελτιώνει αισθητά όχι μόνο την πρόσβαση αλλά και την ποιότητα των αποφάσεων. Και έτσι θα έχουμε ίσες και αποτελεσματικές ε, συνθήκη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η μεγαλύτερη εναρμόνιση μεταξύ των διαφόρων εθνικών συστημάτων είναι πάρα πολύ σημαντικό και εγγράφεται και πάλι σε ένα νέο πολιτικό και νομικό πλαίσιο με τη θέση σε ισχύ της συνθήκης Λισαβόνας. Οι ελάχιστες προδιαγραφές ε, και η σημερινή οδηγία θα πρέπει να αντικατασταθούν από κοινέ προδιαγραφές που είναι πιο φιλόδοξο σχέδιο. Δεν θέλω να σας εξαντλήσω αλλά να θυμίσω τη φιλοσοφία του κειμένου. Η βελτίωση των διαδικασιών στο πρώτο βαθμό εξέταση είναι προ όφελο και των κρατών μελών και των ετούντων άσυλο. Θα πρέπει να είναι ποιοτική η λήψη των αποφάσεων, δηλαδή από τον πρώτο βαθμό, έτσι ώστε οι αρμόδιε αρχέ να παίρνουν ε, γερές, στερέ αποφάσει, να δικαιολογούν τι ανητικέ και έτσι να μειώνεται και ο κίνδυνο ακύρωση του από τι αρχέ στι οποίε προσφεύγουν οι ενδιαφερόμενοι ε, να μειωθούν οι ε, μη ε, βάσιμες ή καταχρηστικές αποφάσεις. Αν θέλετε μπορώ να πω και σε λεπτομέρειες σχολιάζοντας το έγγραφο εργασίας, αλλά θέλησα στην προσέγγιση μου να περιορίσω όσο γίνεται περισσότερο τις δυνατότητες εξαιρέσεων ή παρεκκλήσεων για να μην ξεφεύγουν οι διαδικασίες. Όπως σας είπα, οι εξαιρεσει και πολλοί περιορισμοί που περιλαμβάνονται στο σημερινό κείμενο οδήγησαν όχι μόνο σε ε, αποκλήσεις, αλλά αποκλίνουν και οι δικονομικές εγγυήσεις ε, στα κράτη-μέλη και είναι ε, πολύ, πολλές φορές η κατάσταση αρνητική και καθόλου ικανοποιητική. Αυτά, αγαπητοί συνάδελφοι, όπως και τους τελευταίους μήνες ε, θα είμαι πολύ ε, πρόθυμη να ακούσω ότι έχουν να μου πούν οι σκιώδεις ηγητές. Το έπραξα και στο παρελθόν όπως σας είπα και συμμετείχαν με τρόπο πάρα πολύ δραστήριο και πάρα πολύ επίμονο και ε, επιμελή. Και βέβαια προσβλέπω να ακούσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο, γιατί μπορεί να τηθούν κάποια ερωτήματα ενδεχομένως ως προς αυτά που ακούμε για την αναδιατύπωση του κειμένου ή για το πώς προχωρούν οι συζητήσεις στο Συμβούλιο. Γιατί ακούω, αλλά το βλέπω και στην πρακτική, ότι είναι πάρα πολύ περίπλοκα τα πράγματα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε την κυρία Γκυγιόμ. Κυρία Φλότρ. Σας ευχαριστώ. Όπως ε, θύμισε η εισηγήτρια Σιλβί Γκυγιόμα, Έχουμε συναντηθεί πολλές φορές για να μπορέσουμε να δουλέψουμε πάνω στα διάφορα άρθρα αυτή τη πρόταση. Εγώ θα πρέπει να σας πω πως είμαι πολύ ικανοποιημένη από τα έγγραφο εργασία που μας παρουσιάζει σήμερα. Νομίζω πως ε, δείχνει πραγματικά, ακόμα και αν δεν είναι απόλυτα ε, πλήρε, δείχνει Ποιε είναι οι φαιές ζώνε, ποιε είναι οι μαύρε τρύπε της πρόσβασης στο άσυλο τη σήμερα ημέρα στην Ευρώπη. Υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στι χώρε, αλλά και σταθερά στοιχεία όπως οι συνοριακές περιοχές, όπως ε, το τι συμβαίνει με τους ανήλικους, με τις διάφορες εγγυήσει που υπάρχουν, τις έννοιες ε, του, την έννοια του απορριπταίου αιτήματο ή τις επιτυχημένες διαδικασίες, οι οποίες όμως πολλές φορές δέχονται διάφορες επικρίσεις, γιατί πολλές φορές έχω ακούσει τον Επίτροπο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης ε, να κατακρίνει την ε, καταχρηστική χρήση αυτή της επιταχυμένης διαδικασίας και πιστεύω ότι αυτά που μας ε, καλεί να κάνουμε αυτό το έγγραφο είναι να βασιστούμε σε κοινούς ευρωπαϊκούς κανόνες που θεσπίζουν κάποια βασικά στοιχεία, ότι δηλαδή οποιοδήποτε και οπουδήποτε μπορεί να έχει πρόσβαση σε μια διαδικασία αίτησης για προστασία, μια διαδικασία αξιόπιστη και αυτό σημαίνει κάποιες αλλαγές όπως αυτές που εγγυώνται την νομική στήριξη σε όλη τη διαδικασία, τη διάρκεια μάλλον της διαδικασίας, να, μπορούμε, να μπορεί κανείς να έχει συστηματικά πρόσβαση σε προσφυγή, η οποία να μπορεί να είναι αιρετή, δηλαδή να μην υπάρχει κίνδυνος ε, παραβίασης της αρχής της μη επιστροφής και έπειτα Έχουμε και κάποια θέματα αρχής ε, που δυστυχώς δεν γίνονται σεβαστά σε πολλές ε, χώρες και σε πολλές ε, διοικήσεις που τελικά καταχρώνται του δικαιώματος να λαμβάνουν αποφάσεις που τελικά έχουν όμως πολλές φορές δραματικές συνέπειες για τους ανθρώπους εγώ είμαι ικανοποιημένη λοιπόν από την συνεργασία, από την πρόταση της εισηγήτριας, υποστηρίζω την πρότασή της και σίγουρα τις πολύ ξεκάθαρους στόχους και προθέσεις που περιλαμβάνονται σε αυτό το έγγραφο εργασίας. Νομίζω πως είναι ένα έγγραφο απαραίτητο για την ύπαρξη ενός ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου και είναι απαραίτητο ε, να συμμετέχει και να δεσμευτεί το Συμβούλιο στη διαδικασία οποία μεταρρύθμιση αυτής της οδηγίας, γιατί διαφορετικά θα ήταν τελείως ε, παράλογο να μιλάμε για κοινό ευρωπαϊκό ε, σύστημα ασύλου. Θα πρέπει λοιπόν η μεταρρύθμιση αυτή να συμπεριληφθεί στο πακέτο μεταρρυθμίσεων με στόχο τη θέσπιση ενός κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου που να είναι πραγματικά αξιόπιστο και που θα μπορούμε σε κάθε μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να αγγιηθούμε ένα αποτέλεσμα. Δεν θα πρέπει λοιπόν να μας ξεφύγει αυτή η διαδικασία, αυτή η μεταρρύθμιση, ε, να, γιατί είναι πολύ σημαντικό, όπως σας είπα, στοιχείο για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Μόνικα Όλμαγερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι. Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τη συνάδελφο Σιλβίκη Γιώμ για το έγγραφο εργασία που μας ε, υπέβαλε όπου συμπεριλαμβάνει τα βασικότερα σημεία του προβληματισμού της και μας δίνει και μια εικόνα για το πώς φαντάζεται τη βορεία των πραγμάτων που θα ακολουθήσει τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συμφωνούμε όλοι ότι θέλουμε ελάχιστε προδιαγραφές. Ιδιαίτερα όταν σκέφτομαι ότι θα πρέπει ένας που ζητάει άσυλο να έχει τη δυνατότητα ας πούμε υπηρεσιών διερμηνίας για να καταλαβαίνει ε, τι συμβαίνει και να τον καταλαβαίνουν. Και εκείνη βέβαια χρειάζεται εξήγηση εδώ σε κάποιους ε, ορισμούς. Το πρώτο τι είναι η δωρεάν νομική αρρωγή γιατί χωράει πολλές ερμηνείες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας είπε την περασμένη φορά ότι στην Αυστρία ισχύει ένα σύστημα πάρα πολύ επιτυχές, δηλαδή υπάρχει μια υπηρεσία που παρέχει νομικές συμβουλές. Εγώ έψαξα τι γίνεται στην Αυστρία. Είναι δύο πιλωτικά πειράματα και ακόμα δεν έχουν βγάλει τα συμπεράσματά τους γιατί ακόμα είναι σε λειτουργία. Μετά πήγα στην Αγγλία και ρώτησα τι γίνεται από πλευράς νομικής αρρωγής. Η Αγγλία το απορρίπτει γιατί δεν πήγαν τόσο ρόδινα τα πράγματα όπως μας τα περιέγραψε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σωστό είναι να παρέχονται νομικές συμβουλές για να ξέρει εκείνος που ζητάει άσυλο τι δυνατότητες έχει. Ή αν εμπίπτει σε άλλη κατηγορία μετανάστευσης και να μπορέσει να ζητήσει κάτι άλλο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει Όμω θα πρέπει να είναι πάντα δωρεάν. Εγώ δεν έχω αντίρρηση για νομική συνδρομή. Αλλά αν ε, ο καθένα έχει δωρεάν δικηγόρο και εξαντλεί τα διάφορα στάδια της δικαστικής διαδικασίας που μπορεί να είναι και πέντε από χώρα σε χώρα, αυτό το βρίσκω πάρα πολύ προβληματικό. Χρειάζεται λοιπόν συζήτηση εδώ για να δούμε τι συζητάμε, αν είναι νομικές συμβουλές ή αν είναι σωστό από την πρώτη μέρα, από το πρώτο βήμα της διαδικασίας, καλημέρα σας, ορίστε πάρτε και ένα δωρεάν δικηγόρο. Ε, αυτό φαίνεται κάπως προβληματικό. Εντάξει, το καταλαβαίνω ότι χρειάζεται βοήθεια εκείνο που ζητάει άσυλο. Ε, το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό. Η νομική δεν μπορεί να εξαντλήσει ε, τα διάφορα δικαστικά στάδια μόνος του. Μετά, έχω ερώτηση για τη διαδικασία και την οδηγία αυτή ως προς δυνατότητες κατάχρησης. Η κυρία Φλότρο θα μου πει ότι παντού βλέπω καταχρήσεις. Ε, όχι. Δεν βλέπω παντού καταχρήσεις. Εκείνοι που προσφεύγουν στις χώρες μας ε, θα πρέπει να ε, ε, την χάνουν καλή υποδοχή και να είναι γρήγορε και οι διαδικασίε. Και το καλωσορίζω αυτό και εξ ονόματο του ΕΛΚ. Αλλά τι να κάνουμε, υπάρχουν και καταχρήσει στο δίκαιο του ασύλου και θα πρέπει οι αρχέ και οι υπηρεσίε να έχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίζουν αυτά τα στρεβλά φαινόμενα. Χαίρομαι ιδιαίτερα για το γεγονό ότι θα λαμβάνονται υπόψη ιδιαίτερε ε, συνθήκε ιδιαιτερότητε, α πούμε, ηλικιωμένοι, ε, ανήλικοι, κάποιοι άνθρωποι που έχουν ιδιαίτερα προβλήματα υγεία. Βεβαίω θα πρέπει με αξιοπρέπεια, με ευπρέπεια και με ε, ιατρική περίθαλψη να τους δεχόμαστε. Βεβαίω, δεν διαφωνεί κανεί εδώ. Δυσκολεύουν τα πράγματα όταν θα πρέπει να απαντήσουμε στο τι θα κάνουμε, πώς θα αποτρέψουμε δηλαδή κάποιοι δουλέμποροι και εγκληματίες προσπαθούν να χειραγωγήσουν οικογένειες για να δώσουν πολλά λεφτά ας πούμε, για τη διακίνηση ανηλίκων και να φέρνουν σε μας ε, ανηλίκους ε, να υποφέρουν στον δρόμο τα πάνδυνα με, με τέτοια ψυχικά τραύματα και άλλα που, ας πούμε, που δεν έρχονται και στις χώρες μας πάντα αλλά ας πούμε ότι φτάνουν, μετά δεν μπορούν ποτέ να ξεπεράσουν αυτά τα τραύματα. Δηλαδή, εμείς έχουμε καλές προθέσεις, καλές ρυθμίσεις, αλλά δεν θα πρέπει ε, να ε, αφήνουμε παραθυράκια σε δουλεμπόρους, σε αυτές τις κατηγορίες ακριβώς να ε, εγκληματούν. Βεβαίως, τα παιδιά και οι ανήλικοι θα πρέπει να έχουν πρόσβαση και σε μόρφωση και σε εκπαίδευση βεβαίως. Και καλό είναι να πηγαίνουν σχολείο. Είτε αυτό είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση είτε είναι στις χώρες τους. Είναι πάντα σωστό για τα παιδιά η εκπαίδευση και η μόρφωση δεν έχει βλάψει ποτέ κανένα. Τώρα το θέμα της εξαφάνισης των ε, ε, προσώπων αυτών. Δηλαδή, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπει ότι αν αυτοί εξαφανιστούν και πέσουν στην παρανομία, να μην μπορεί να κλείσει η διαδικασία. Δηλαδή, να έχει τη δυνατότητα, δηλαδή, όποιος το κάνει αυτό, να μην χάνει την ε, ε, το φάκελό του στο, στην υποβολή ασύλου να εξακολουθεί να ισχύει. Γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει. Δεν με βρίσκει σύμφωνη αυτό. Ε, και ε, αμφιβάλλουν και πολλοί νομικοί. Αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εννοεί αυτό που λέει, ότι δεν θέλει να σπρώχνει στου ανθρώπου αυτού στην παρανομία, τότε να δώσει τα κράτη-μέλη και τα απαραίτητα εργαλεία που χρειάζονται για να το αντιμετωπίσουν η ταχεία διαδικασία είναι κάτι που βρίσκω εγώ πάρα πολύ προβληματικό επίσης. Υπάρχουν κάποιες υποχρεώσεις ε, και συνεργασίες. τους δίνουμε την εγγύση ότι έχουν ασφαλή διαμονή θα πρέπει όμως να μας λέει ο ενδιαφερόμενος και το πραγματικό του όνομα και την πατρίδα του και να βοηθάει λίγο και εκείνο να συνεργάζεται. Γιατί θέλει οπωσδήποτε άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν δεν συνεργάζεται ο ενδιαφερόμενος δεν μπορούμε να έχουμε επιταχυμένες διαδικασίες και πάλι το βρίσκω αυτό προβληματικό. Δηλαδή επιβραβεύεται κάποιο που μετέρχεται αυτό το μέσο. Και χαίρομαι μεν για το γεγονό ότι θέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να περιορίσει το χρόνο τη διαδικασία σε ένα εξάμεινο, αλλά καταλαβαίνουμε και ξέρουμε πόσα εμπόδια μπορεί κανεί που δεν ενδιαφέρεται ε, να προχωρήσει γρήγορα να, να, να ορθώσει εμπόδια μέσα σε αυτό το εξάμεινο. Και μετά θα έρχονται τα κράτη-μέλη να δικαιολογούν γιατί δεν τήρησαν το εξάμεινο. Γιατί είμαι σίγουρη ότι δεν πρόκειται να το τήρησουν. Αφήστε δε που προσφέρεται αυτό για την ε, δημιουργία εμποδίων προς κομμάτων. Χρειάζεται συζήτηση αυτό για όλα αυτά τα θέματα. Είμαι υπέρ, επαναλαμβάνω, των ταχαίων διαδικασιών, αλλά θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν και τα κράτη-μέλη αυτό και να υποχρεώνουν τους ετούντες ασύλου έτσι, ε, ε, μια στοιχειώδη συνεργασία να τη δείχνουν. Τώρα υπάρχουν και πραγματικά ψυχικά τραύματα και θα πρέπει να εξασφαλίζεται και ιατρική περίθαλψη ε, στον ενδιαφερόμενο υποστήριξη για να μπορεί να βοηθάει και εκείνος στις αρχές, αλλά αυτό να μην γίνει εμπόδιο για ε, επαναπροώθηση ή απέλαση ή οτιδήποτε τη διαδικασία. Συμπέρασμα, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα θέλει πραγματικά ε, ένα χώρο προστασίας για εκείνου που διώκονται, αλλά να είναι και καλύτερες οι υπηρεσίες προσφυγής Δηλαδή, πολλοί από εκείνους που ζητούν άσυλο έχουν έρθει παράνομα στις χώρες μας, μέσω δικτύων ε, δουλεμπόρων ε, και ε, υπηρεσίε τι οποίε θα μπορούσαν να αποτείνονται εκτό τη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχουν σήμερα. Είναι πολύ ελάχιστε. Θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα κάποιο που θέλει να έρθει στην Ένωση να απευθυνθεί σε μια υπηρεσία εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση εφόσον διώκεται για να βοηθηθεί. Να έρθει στι χώρε μα, δεν λέω. Τώρα κάποιοι που θέλουν απλώς μια καλύτερη ζωή και το καταλαβαίνουμε όλοι, αλλά δεν μπορούμε να σώσουμε τον κόσμο όλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εν πάση περιπτώσει να τους δίνουμε τη δυνατότητα να ενημερώνονται πριν πέφτουν σε χέρια ε, δουλεμπόρων, εγκληματιών και ζούμε καταστάσεις όπως αυτές που άκουσα την περασμένη εβδομάδα που μια τέτοια συμμορία παράτησε στην έρημο ανθρώπους που τους είχε προηγουμένως γδίσει οικονομικά και τους άφησε να πεθάνουν από τη δίψα. Ευχαριστώ και τη Σιλβί Γκυγιό που έκανε πολλές συνεδριάσεις με τους γεωδησηγητές για να μας ακούσει και εμά και παρακαλώ για κάποιες διευκρινήσεις σε ορισμένους τομείς. Γιατί ε, ε, παραμένουν πολλά εμπόδια για τη διαδικασία και το εξάμεινο είναι πολύ δύσκολο. Χρειάζεται αυτό συζήτηση. Πώς θα αντιμετωπιστούν φαινόμενα κατάχρησης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Το λόγο τώρα έχει ο κύριος Μπρόνς. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ξέρω ποια αναλογία των ετών των άσυλο έχει έρθει άμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τη χώρα από την οποία ξεκίνησε, λόγω της υποτιθέμενης δίωξής τους. Και ποιο ποσοστό έχει περάσει από ασφαλείς χώρες. ότι από αυτούς μπορεί όντως να είναι γνήσιοι για τον άσυλο ακόμα και αν αυτοί που περνάνε από ασφαλείς χώρες αρχικά ε, ε, αναζητούσαν άσυλο από τη στιγμή που έχουν ε, παρακάμψει μία μόνη ασφαλή χώρα στην ουσία μετατρέπονται σε παράνομους οικονομικούς μετανάστες. Το να τους αντιμετωπίζουμε ως τον άσυλο είναι άδικο για αυτούς που πραγματικά ζητούν προστασία αποδίωξη στη χώρα τους. Ευχαριστώ. κυρία Βέμπερ. Ευχαριστώ. Καταρχάς, θα ήθελα να σας ζητήσω συγγνώμη εξ ονόματος της συναδέλφου Νάντια Χέτς που είναι σκιώδης ηγήτρια των φιλελευθέρων ε, αλλά σήμερα έχει μια ανηλμένη υποχρέωση και δεν μπόρεσε να παρευρεθεί. Να σας πω ποια είναι η θέση της ομάδας μας των φιλελευθέρων για το θέμα αυτό, αλλά γενικότερα για το πακέτο του ασύλου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για τη σημερινή παρουσίαση και το έγγραφο εργασίας που μας υπέβαλε. Η ομάδα μας θεωρεί ότι θα πρέπει να υιοθετήσουμε μια κοινή θέση όλοι μας απέναντι στο θέμα του ασύλου. Ορισμένα από τα στοιχεία αυτά καταλαβαίνουμε ότι χρειάζονται ε, διαφορετική μεταβατική περίοδο σε κάθε χώρα μέχρι να εφαρμοστούν, αλλά είναι μια κοινή προσέγγιση για όλο το πακέτο. Ξέρουμε ότι το Συμβούλιο δεν συμφωνεί. Ε, πάντα σε αυτά που λέμε. Πέρα από τις ιδεολογίες λοιπόν που έχουμε στο Κοινοβούλιο θα πρέπει να υπάρξει μια κρίσιμη μάζα συναδέλφων, ένα ικανό ε, ποσοστό, ε, ικανός αριθμός που να θέλουν να καταλήξουν στην κοινή προσέγγιση. Σε ό,τι αφορά το έγγραφο συγκεκριμένα της κυρίας Γκυγιόμ, την ευχαριστώ για τις ερωτήσεις που έθεσε για διάφορα θέματα. που βρίσκονται στην πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εμείς οι φιλελεύθεροι θεωρούμε ότι είναι φυσιολογικό να υπάρχουν προδιαγραφές, έστω και ελάχιστε προδιαγραφές, ναι, σε πολλούς τομείς. Το δικαίωμα στη δωρεάν ε, παροχή νομικής ε, υποστήριξης ή ε, προσφυγή σε ανώτερο βαθμό δικαιοσύνη. Όλα αυτά θα πρέπει να τα λύσουμε. Τι γίνεται με τους ασυνόδευτους ανηλίκους και επίσης τι γίνεται με τις περίφημες έννοιες της ασφαλούς χώρας, ασφαλής χώρα ε, προέλευσης, ασφαλής χώρα διέλευσης, ασφαλής ευρωπαϊκή χώρα, ασφαλής τρίτη χώρα. Να καταλάβουμε τι είναι όλα αυτά για να μην έχουμε συγχύσεις ε, όταν κληθούμε να εφαρμόσουμε το κείμενο. Δεν χρειάζεται να το υπογραμμίσω, θα το κάνω όμως, γιατί πιστεύω ότι αν δεν κινηθεί ταχύτατα το Κοινοβούλιο να κάνει ένα κείμενο και να το υποβάλει στο Συμβούλιο για να συμφωνήσει με τις προτάσεις μας στο Συμβούλιο, δεν τα κάνουμε όλα αυτά λοιπόν και εάν δεν καταφέρουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να έχουμε κοινή αντιμετώπιση, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι τελικά τα κράτη-μέλη θα κάνουν εκείνα ό,τι επιθυμούν και δεν θα μας λάβουν υπόψη. Δεν το θέλουμε εμείς αυτό. Καταλαβαίνω πολύ καλά ότι υπάρχουν ε, διαφορετικά συμφέροντα στα διαφοροκρατή μέλη, γιατί δεν πλήττονται κατά τον ίδιο τρόπο όλες οι χώρες. Αυτό είναι προφανές για όλους, αλλά θα πρέπει να καταλάβουμε ταυτόχρονα ότι και οι άνθρωποι αυτοί είναι άνθρωποι, σαν και εμά, που για διάφορους λόγους ασφαλείας ή κινδυνεύει η ζωή τους ε, καταφεύγουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είναι λογικό και επόμενο και φυσικό τα παράπονά τους και ε, τα αιτήματά τους να γίνονται ακουστά αν μη τι άλλο και σεβαστά. Η έκθεση λοιπόν θα πρέπει το συντομότερο να κατατεθεί από την κυρία Κιγιόμ για να μπορέσουμε και εμείς να ανταποκριθούμε στην αρχική μας επιθυμία να εγκριθεί μέχρι το 2012 αυτή η οδηγία. Ευχαριστώ. Μάλιστα, ευχαριστώ κύριε Μπουζούτιλ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν να, ευχαριστώ, να, να, ευχηθώ χρόνια πολλά στον ε, Δεμέρα που είναι η γενέθλιά του σήμερα. Αλλά δεν τον βλέπω πια στην αίθουσα. Μέχρι να πάρω το μικρόφωνο ε, εξαφανίστη. Μπάς περιπτώσει θα ξανάλθει. Τις καλύτερες ευχές μου λοιπόν για την γενέθλιά του. Στην ε, παρέμβασή μου θα ήθελα να βασικά να στηρίξω τα όσα είπε η συνάδελφος Μόνικα Χολμάγερ Εγώ προέρχομαι από μια χώρα που είναι τελείω διαφορετική όσον αφορά την πραγματικότητα της ε, χώρας της Μόνικας. Ωστόσο, συμμερίζομαι πολλές από τις παρατηρήσεις που έκανε. Να αρχίσω λέγοντας ότι και εγώ συμφωνώ ότι πρέπει η νομοθεσία να είναι ξεκάθαρη για αυτό το θέμα και ότι η νομοθεσία αυτή θα πρέπει καταρχήν να μας, να μας βοηθήσει επισήμως να μπορέσουμε να ξεχωρίσουμε αυτούς που πραγματικά χρειάζονται διεθνή προστασία από αυτούς που δεν χρειάζονται τέτοιο πράγμα. Γιατί υπάρχει διαφοροποίηση και πρέπει να γίνει προς όφελος όλων αυτών που όντως χρειάζονται προστασία. Εάν δεν το κάνουμε αυτό, θα δημιουργήσουμε μια νομοθεσία η οποία θα είναι μόνο βάρος, θα δίνει λαβή για κατάχρηση και αυτό βέβαια εις βάρος των ανθρώπων που πραγματικά και γνήσια χρειάζονται προστασία. Γιατί οι πραγματικές περιπτώσεις θα πνιγούν μέσα στους χήμαρους καταχρηστικών περιπτώσεων. Η, ελεύθερη, η δωρεάν ας πούμε, νομική βοήθεια αλλά και η χρήση της επιταχυμένης μεθοριακής διαδικασίας γίνεται όλα ένα και πιο δύσκολη σύμφωνα με αυτήν εδώ την πρόταση. Και να ολοκληρώσω λέγοντας μόνο το εξής Όλα είναι ωραία και καλά εδώ για μας. Εδώ εμεί ε, μπορούμε να ακολουθήσουμε μια διαδικασία τελείω τυπική, να αυξήσουμε τα στάνταρ, να εισάγουμε περισσότερα δικαιώματα και είναι πολύ θετικό να αυξάνονται τα δικαιώματα. Ποιο θα ήταν κατά κάτι τέτοιο. Ωστόσο πρέπει να προσέξουμε να μην είμαστε τελείω άσχετοι από την πραγματικότητα από το τι συμβαίνει επί τόπου. Και υπάρχουν πολλά κράτη-μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εγώ προέρχομαι από ένα από, ένα από αυτά τα μέλη και βλέπω και τον συνάδελφο Σταύρο Λαμπρινίδη που είναι εδώ και είναι από την Ελλάδα. Υπάρχουν λοιπόν πολλά κράτη-μέλη που αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλες δυσκολίες με την νομοθεσία που ισχύει σήμερα. Πόσο μάλλον αν βάλουμε νέα νομοθεσία που να αυξάνει ακόμα περισσότερο τι δυσκολίες. Ε, γιατί, γι' αυτό νομίζω πω πραγματικά θα πρέπει να βοηθηθούν αυτά τα κράτη-μέλη. Καταρχήν να συμμορφωθούν με τα στάνταρ που ισχύουν σήμερα. Είναι ήδη εξαιρετικά δύσκολο για μας. Στην ουσία έχουν μείνει, έχουν μείνει τα κράτη αυτά μόνα τους και αντιμετωπίζουν ε, την, ε, όλη την πόρα και αυτή τη στιγμή αυτό που κάνουμε είναι να μετακινούμε το τέρμα. Ε, αλλάζουν τους κανόνες του παιχνιδιού. Ε, είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Προσέξτε συνάδελφοι, γιατί δεν πρέπει να απομακρυνθούμε, όπως σας είπα, από την πραγματικότητα που ισχύει επί τόπου. Ναι, χρειαζόμαστε νομοθεσία, ναι, χρειαζόμαστε καλά ε, και υψηλέ προδιαγραφές, γιατί όπως και η Νάτ Βέμπερ, εδώ έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους, αλλά όλα αυτά θα πρέπει να είναι ρεαλιστικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ε, να ευχηθώ και εγώ εξ ονόματο όλων μα ε, στον Δίας Δεμέρα χρόνια πολλά, είναι τα γενέθλιά του. Πριν το έκανε ο Σέμον Μουζουτήλ πριν να μπει στην αίθουσα. Τα 80 κλείνει, αλλά δεν του φαίνεται καθόλου. Το λόγο τώρα έχει ο κύριος Φαντεστούπα. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν, κυρία Γκυγιό Ευχαριστώ την Σκιώδη Συγκήτρια, ε, αλλά δεν είμαι βέβαιος ότι έγιναν πολλές διαβουλεύσεις. Ας πούμε, η κυρία Κικιόμ δεν έλαβε υπόψη τους εκλογείς του κόμματος της Ελευθερίας στις, των κάτω χωρών και ήθελα πραγματικά να αντιδράσει σε αυτά που τους είπα. Εμείς είμαστε αντίθετοι ενός συστήματος ασύλου σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ήθελα να αναφέρω κάποια σημεία ως προς την ουσία. Ας πούμε, υιοθετήθηκε η αρχή της επικουρικότητας, αλλά δεν είναι πιστική και σίγουρα ορισμένα κομμάτια αυτού του συστήματος δεν είναι καθόλου πιστικά. Και επιπλέον αυτά που είπε η Κομισιόν, ότι αυτή η μεταρρύθμιση θα διασφαλίσει, λέει, καλύτερη συνοχή στην πολιτική ασύλου, μια απλοποίηση της διαδικασίας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καλύτερη λήψη αποφάσεων που επιτρέπει να αποφεύγονται οι καταχρήσεις. Και γι' αυτό ρωτώ το καλύτερη λήψη αποφάσεων, τι θα πει αυτό, καλύτερες αποφάσεις για τους ετούντε άσυλο ή για τα κράτη-μέλη που είναι οι παραλήπτες των τον Και έπειτα μου λέτε για αποφυγή των καταχρήσεων αν υιοθετηθεί μια απλοποίηση της διαδικασίας. Πραγματικά, ειλικρινά, πολύ αμφιβάλλω αν θα συμβεί κάτι τέτοιο. Τα κράτη-μέλη θέλουν να έχουν προδιαγραφές ευνοϊκές για αυτές τις διαδικασίες και διαδικασίες που να λειτουργούν ε, ε, εύρυθμα. Ναι, αλλά για ποιον, επαναλαμβάνω. Και μετά κάνουμε λόγο για τους ετούντες άσυλο που φτάνουν σε μια χώρα και που μετά παραμένουν και γίνονται λαθρομετανάστες. Πώς γίνεται αυτό και πώς ένα κράτος μέλος μπορεί να αποδείξει ότι κάποιος που τον άσυλο τελικά μετατρέπει σε παράνομο μετανάστη. Και έπειτα για τον τραυματισμό της αναχώρησης τελικά οι τοπικοί δικαστές δεν είναι αυτοί που θα πρέπει να δράσουν και όχι ε, το κοινοτικό επίπεδο. Δηλαδή, ναι, μπορούμε να δώσουμε κάποιες οδηγίε στου δικαστέ, ξεκάθαρα. Και αλλαγή της ορολογίας επίσης. Και εδώ θέλω να επανέλθω, γιατί νομίζω πώ είναι τη ορολογία επίση. και εδω θελω να επανελθω γιατι νομιζω πω ειναι χαρακτηριστικο των όσων κάνουμε ανέκαθεν. Δίνουμε άλλο όνομα στο ίδιο πράγμα. Και δεν μιλάμε τώρα για τον τάσυλο, μιλάμε για ένα αίτημα ασύλου, που μετατρέπεται σε αίτημα διεθνού προστασία. Πραγματικά αυτά όλα είναι αξιοθρύνητα. Δίνουν μια εικόνα για την πραγματικότητα πραγματικότητα που δεν αντιστοιχεί καθόλου τελικά στην πραγματικότητα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να επανέλθω σε κάποια βασικά σημεία αυτού που συζητάμε είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη για όλη την διαδικασία να καταλήξουμε σε κοινά πρότυπο για μια κοινή διαδικασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό πρέπει να διασφαλιστεί με κάποιο τρόπο. Σαφώ η κατάσταση σε κάθε κράτο μέλο είναι διαφορετική, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να υπάρχουν κάποια πρότυπα. σα ίσα είναι απαραίτητα και θα πρέπει να προσέξουμε και να υπάρξει και μια αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών. πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα περισσότερο. Όσον αφορά τώρα τη διαδικασία των έξι μηνών, θα πρέπει να είναι σαφές το εξής. θα πρέπει να συνεργάζεται και αυτός που καταθέτει την αίτηση ασύλου. Από εκεί και πέρα το πόσο θα διαρκέσει μια διαδικασία εξαρτάται και από το προσωπικό το οποίο είναι στη διάθεση ε, μιας υπηρεσίας και από την ποιότητα του προσωπικού που ασχολείται με τη διαδικασία και τις ε, απαραίτητες ε, διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο πρόσφυγας που κάνει αίτηση ασύλου. και δεν είναι βασικά οικονομικά τα προβλήματα. Ως Ευρωπαϊκή Ένωση πάντα είμαστε πάρα πολύ πρόθυμοι να ε, συζητάμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα πανταχού της γης. Άρα θα πρέπει να αναρωτηθούμε και εμείς πώς τηρούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και να μην το ξεπουλάμε κόψω χρονιά, να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προστατεύουμε εκείνους που πραγματικά χρειάζονται προστασία. Και να ξεκαθαρίζουν τα πράγματα. Και το θέμα της εξαφάνισης, όταν κάποιος δηλώνεται και μετά χάνεται στην παρανομία. Και αυτό θα πρέπει να το εξετάσουμε. Το έχω ξαναπεί εδώ στην Επιτροπή μας. Ή το άλλο, το θέμα το περίφημο των ασφαλών χωρών διέλευση. Και αυτό πρέπει να το ξανασυζητήσουμε εδώ στην Επιτροπή μας πάρα πολύ εντατικά, γιατί καμιά φορά έχω την εντύπωση ότι αν συνεχίσουμε έτσι τότε Κάθε χώρα της Ιφιλίου θα ονομάζεται ασφαλής χώρα διέλευσης. Και εντάξει. Επίσης παραβλέπουμε το γεγονός ότι και η αφετηρία από την οποία κινούν οι πρόσφυγες είναι διαφορετική. Γιατί μια χώρα που μπορεί να είναι ασφαλής, μια τρίτη χώρα για κάποιον πρόσφυγα, μπορεί να μην είναι ασφαλής για έναν άλλον. Έτσι και ως Ευρωπαϊκή Ένωση θέλουμε να είμαστε και υπόδειγμα λέμε για την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να μην χανόμαστε στις ε, λεπτομέρειες ε, της συζήτησης με τρόπο μικρόψυχο. Ευχαριστώ κύριε Ρομέρο Λόπες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι σε αυτή την οδηγία συζητάμε τη διαδικασία και τους ελάχιστους κανόνες ώστε τα κρατη μελη να πλουστεύσουν τη διαδικασία και να εξοικονομήσουν και κάποιους πόρους. Είμαι πεπισμένη ότι όλες οι πολιτικές ομάδες συμφωνούμε εδώ στο Κοινοβούλιο Συμφωνούμε ως προς το γεγονός ότι οι καταχρήσεις δεν επιτρέπουν να ε, ακολουθούμε τις σωστές διαδικασίες για αυτούς που πραγματικά είναι τούντες άσυλο και χρειάζονται διεθνή προστασία. Αυτό που δεν μπορούμε να κάνουμε είναι να χρησιμοποιήσουμε αυτή την οδηγία για να συζητήσουμε πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με το ζήτημα που συζητάμε. Δηλαδή, δεν μπορούμε να μιλάμε για καταχρήσεις που σχετίζονται με ε, Διότι αυτός ο οποίος κάνει αίτηση ασύλου ή ζητά διεθνή προστασία, εάν επιπλέον είναι ε, και θύμα δουλεμπορίου, είναι ουσιαστικά διπλά θύμα. Και, επειδή, και δεν μπορούμε να σκεφτούμε ότι επειδή υπήρξε θύμα δηλεμπορίας δεν δικαιούται ασύλου όταν ταυτόχρονα έχει βρεθεί σε μια κατάσταση η οποία αποτελεί τραγωδία για τη χώρα του. Δεν μπορούμε να αναμειγνύουμε τα δύο πράγματα διότι δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ των και ε, ε, πόσο μάλλον εάν πρόκειται για κάποιο άτομο το οποίο είναι ανήλικο. Εάν κάποιο είναι ανήλικο είναι ακόμα μεγαλύτερη ανάγκη προστασία. Αυτό που κάνει αίτηση ασύλου και χρειάζεται διεθνή προστασία, εάν πραγματικά την αξίζει, ανεξάρτητα από το αν υπήρξε ε, θύμα δουλεμπόρων, την αξίζει. Εδώ συζητάμε τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθούν τα κράτη-μέλη. Δεν, ακολουθού, δεν συζητάμε άλλο θέμα. Το, το άλλο ζήτημα θα το συζητήσουμε αργότερα. Εάν λοιπόν το παρουσιάσουμε αυτό ως πρόσχημα για να προασπίσουμε μια κατάσταση η οποία στην πραγματικότητα δεν είναι πολύ σαφής και δεν θα πρέπει να αποφασίσουμε για να δούμε, το χρησιμοποιήσουμε σαν αντικείμενο για να δούμε αν γίνεται κατάχρηση, ε, τότε ε, δεν έχουμε στεναρά επιχειρήματα. Διότι δεν πρέπει να αναμειγνύουμε τη διαδικασία και την κατάσταση που έχουμε σε κάθε κράτος μέλος προκειμένου να πλουστεύσουμε τη διαδικασία με το δουλεμπόριο είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Και όταν συζητάμε για δουλεμπόριο, συζητάμε για ένα άλλο ζήτημα το οποίο δεν έχει καμία σχέση. Ορισμένε φορές έχουμε άτομα τα οποία έχουν υπάρξει χρήματα και στις δύο περιπτώσεις. Έχουμε άλλες δύο παρεμβάσεις. Η κυρία Λάτφορτ. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε και την κυρία Γκυγιόμ για το πολύ χρήσιμο έγγραφο εργασία τη. Η Βρετανική κυβέρνηση ενημέρωσε προσφάτως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι αναστέλει τις επιστροφές στην Ελλάδα προσωρινά βάσει του κανονισμού του Δουβλίνου, διότι έχουμε 1.300 ετούντες οι οποίοι ακόμα βρίσκονται υπό διαδικασία έρευνα στα βρετανικά δικαστήρια και εκτιμάται ότι σε κάποιες περιπτώσεις θα έχουμε δύο χρόνια ε, συζητήσεων ε, υπάρχουν άτομα τα οποία φυσικά δεν είναι όλες οι περιπτώσεις αυτές αλλά κάποιοι εξ αυτών αρνούνται να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Το Ηνωμένο Βασίλειο λοιπόν έχει αποφασίσει να ασχοληθεί προσωπικώ με, την, με τις αιτήσει αυτές και να μην χρησιμοποιήσει το σύστημα του Δουβλίνου. Και εδώ έρχονται πολλές σκέψει. Πρώτον, Εγώ υποστηρίζω εδώ και πάρα πολύ καιρό τις ε, διαδικασίες ασύλου και θέλω να υπάρχουν υψηλές προδιαγραφές, να έχουμε ταύτιση με το διεθνές δίκαιο για να γίνεται ο κατάλληλος έλεγχος ε, για όλους όσους καταθέτουν αίτηση και επίσης να προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα πρέπει να αρνούμαστε προστασία σε οποιονδήποτε τη δικαιούται. Ταυτόχρονα βέβαια θα πρέπει να έχουμε αποτελεσματικές διαδικασίες και ως προς το ε, ε κόστος και κάτι το οποίο συνδέεται και με τους δύο στόχους είναι να υπάρχει και δημόσια υποστήριξη για το σύστημα του ασύλου. Και φυσικά υπάρχουν συνεχείς πιέσεις για τους τρεις αυτούς στόχους. αυτό το οποίο θα πρέπει να περνάει τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας ω προ το κόστο και της αποδοτικότητα είναι οι υψηλέ προδιαγραφές. Διότι αν υπορφαρτώσει κάποιο το σύστημα δεν θα έχει ε, αποφάσει υψηλή ποιότητας. Που θα μας οδηγούν και σε επιτυχή αποτελέσματα. Ω αρχή λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλη υποστήριξη προ του ετώντε, να γίνονται πολύ καλέ ε, προσωπικέ συνεντεύξει. κάτι το οποίο στη συνέχεια ε, λογικά θα δημιουργήσει και κάποιες καθυστερήσεις στο σύστημα, διότι εξαρτώνται από αυτές τις συνεδράσεις, αλλά θα μας επιτρέψει να προσπίσουμε τις αρχικές μας αποφάσεις καλύτερα, ότι θα είναι αποφάσεις οι οποίε θα έχουν ληφθεί ε, με κατάλληλη προετοιμασία, εάν υπάρξει θέμα έφεσης. Δεν ξέρω βέβαια για ποιον ακριβώς λόγο έλαβε αυτή την απόφαση το Ηνωμένο Βασίλειο και δεν θέλω να την υπερασπιστώ απόλυτα, αλλά ε, δεν θα πρέπει να χάσουμε και επαφή με την πραγματικότητα. Αφενός ε, πρέπει να είμαστε φιλόδεξοι σε επίπεδο νομοθεσίας, αλλά θα πρέπει ταυτόχρονα να γνωρίζουμε και πού βρισκόμαστε στην εφαρμογή του πρώτου γύρου της Οδηγίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα στην εφαρμογή και συνεπώς δεν θα πρέπει να είμαστε υπερφιλόδοξοι, διότι το καλύτερο είναι ο εχθρός του καλού το καλό απαιτεί κάθε κράτος μέλος να έχει ένα κατάλληλο σύστημα ε, αποφάσεων για το άσυλο, για το ποιος δικαιούται άσυλο και δυστυχώς αυτό αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Δεν ε, κατηγορώ κανέναν, ξέρω ότι υπάρχουν συγκεκριμένες πιέσεις σε κάποιες χώρες, αλλά γνωρίζω ότι υπάρχουν και κάποιες πρακτικές πτυχές οι οποίες πρέπει να υλοποιηθούν. Υπάρχει το νέο γραφείο υποστήριξης ασύλου, υπάρχει πολύ περισσότερη ε, εκπαίδευση και συνεργασία και θα πρέπει να προσδώσουμε αντίστοιχο βάρος και στην πρακτική εφαρμογή και την πρακτική βελτίωση όσο βάρος δίνουμε και στην ε, απόφαση των νομοθετικών μέτρων. Δεν λέω δηλαδή να χάσουμε το στόχο μας και να ξεχάσουμε τις αποτελεσματικές διαδικασίες υψηλής ποιότητας, αλλά να μην πάμε και προς την τελείως αντίστοιχη, αντίθετη κατεύθυνση. Ένα κοινό σύστημα ασύλου μέχρι το 2012, ας είμαστε ρεαλιστές, δεν πρόκειται να υπάρξει. Να διασφαλίσουμε τουλάχιστον ότι κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε ε, επιτόπου και ε, να μην δίνουμε ουτοπικές προσδοκίες ε, για πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να καταφέρουμε. Ναι, και εγώ θέλω υψηλή ποιότητα ε, και εγώ θέλω να έχουμε ένα εύρωστο σύστημα ασύλου, αλλά δεν νομίζω ότι στα επόμενα δύο χρόνια θα το καταφέρουμε. Κύριε Ολμαγερ, ήθελα μόνο πολύ σύντομα, γιατί αναφέρθηκε σε μένα συνάδελφος, Ε, το 1990 η Γερμανία αναγκάστηκε από τα πράγματα να αποκομίσει μεγάλες εμπειρίες από τις ε, οργανωμένες πύρες δουλεμπόρων. Έχουμε γίνει εμπειρογνώμονες περίπου. Και άλλαξαν ε, οι διαδικασίες και στη Γερμανία ακριβώς τότε. Ιδιαίτερες κατηγορίες, ιδιαίτερες ομάδες, αν τη χάνουν προστασίας, τότε οι δουλέμποροι προσπαθούν να στρέφονται ακριβώς στοχευμένα σε αυτές τις ομάδες και να φέρνουν περισσότερους ε, από τις ομάδες αυτές στα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να προστατεύουμε τους ανθρώπους. Πρέπει. Αλλά να σκεφτούμε πώς είναι οι μηχανισμοί και πώς θα τους αξιοποιήσουμε με τρόπο λογικό για να μην είναι και κίνητρο επιπλέον και δέλεαρ για περισσότερο εμπόριο παιδιών ενώ εμείς θέλαμε αρχικά να προστατεύουμε τους ανηλίκους καλύτερα. Γι' αυτό λέω ότι χρειάζεται διαφορετική, διαφοροποιημένη προσέγγιση με ρεαλισμό, γιατί δυστυχώς έχουμε ζήσει αυτές τις εμπειρίες και δεν ήταν πάρα πολύ θετικές σε κάποιους τομείς. Τώρα, σε μια άλλη θεματική ενότητα, αγαπητή κυρία Ζήπελ, να μην παίζουν τα οικονομικά μεγάλο ρόλο. Και εδώ είμαι ρεαλίστρια. Μπορούμε να επιθυμούμε πολλά αλλά συμφωνώ με την κυρία Λάτφορκα κάπου θα πρέπει να δείχνουμε και ένα ρεαλισμό. Βεβαίω θα πρέπει οι διοκόμενοι να προστατεύονται όσο γίνεται και όσο μπορούμε και είμαστε και φιλεύσπλαχνοι και ό,τι άλλο θέλετε. Αλλά Υπάρχουν κύματα ανθρώπων που έρχονται για διαφορετικούς λόγους στις χώρες μας και αυτό είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα και είναι πολύ δύσκολο για εκείνους που διώκονται ακριβώς να κάνουν τη φωνή τους να ακουστεί που είναι διαφορετική από τη μεγάλη μάζα των, διο... των μη διοκόμενων που έρχονται από άλλα κριτήρια. Δεν είναι μόνο ποσοτικά, είναι και ποιοτικά τα προβλήματα θα πρέπει να έχουμε ένα σύστημα ρεαλιστικό που να διαφοροποιεί τις καταστάσεις με πιο ταχύες διαδικασίες, αλλά όσο γίνεται να αποφεύγεται η κατάχρηση. Να ανοιχνεύεται κιόλας η κατάχρηση. Και να δίνουμε στους ανθρώπους μια ρεαλιστική προοπτική. Και για εκείνους που θέλουν να έρθουν για άλλους λόγους Το θέμα της εξαφάνισης στην παρανομία. Δεν το καταλαβαίνω πραγματικά αυτό που λέτε. Σε μια χώρα όπου υπάρχουν αξιοπρεπείς ελάχιστες προδιαγραφές δεν έχει κανένας λόγο να εξαφανιστεί. Γιατί υπάρχει διαδικασία, είναι δεδομένη, έχει την πορεία της, γιατί να χαθεί ο άλλος. Εγώ δεν θέλω να κατηγορήσω καμία χώρα. Και κυρία Λάτφορτ, προς ενημέρωσή σας, η Γερμανία δεν στέλνει στην Ελλάδα όπως και η Αγγλία πίσω. Ε, έχουμε στείλει όμως πολλούς ε, υπαλλήλους από τη Βαβαρία στην Ελλάδα για συνεργασία και για βοήθεια ε, στην διεκπαιρέωση των φακέλων και των περιπτώσεων. Καλό είναι λοιπόν να βοηθούμε και διοικητικά τις διάφορες υπηρεσίες και τις διάφορες αρχές που το έχουν ανάγκη. Αλλά μια χώρα πραγματικά αντιμετωπίζει ακραίες καταστάσεις θα πρέπει να σκεφτούμε πρακτικά πιο γρήγορα να βοηθούμε ένα τον άλλο και στην ανταλλαγή ε, ετούντων ασύλ από ό,τι στο παρελθόν. Εγώ σε καμία περίπτωση δεν ζητώ να ανοίξει το, η Ευρώπη, να γίνει φρούριο η Ευρώπη. Αλλά αν θέλουμε να βοηθήσουμε πραγματικά τους ανθρώπους που διώκονται, να έχουμε σωστές διαδικασίες, σωστά συστήματα και να μπορούν και τα εμελήματά τους να γίνονται ακουστά. Και να μην χάνονται εκείνοι ε, στους ε, δεδάλους της ε, διαδικασίας. Έχει ζητήσει το λόγο ο κύριος Λαμπρινίδης και μετά θα δώσουμε το λόγο στο Συμβούλιο γιατί έχουμε καθυστέρηση. Uh, πολύ σύντομα θα ήθελα να πω τα εξή. Σαφώς, κατά εμέ, όλο αυτό το πράγμα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ε, σύνολο, ένα πακέτο. Και είναι πολύ σημαντικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και δυστυχώ το Κοινοβούλιο θα πρέπει να είναι αυτό που θα το κάνει, διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο δεν το κάνουν, να σημειώσει πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει ένας μόνιμος μηχανισμός αλληλεγγύης για τα κράτη-μέλη που λαμβάνουν τον μεγαλύτερο αριθμό αιτήσεων ασύλου. Το λέω αυτό διότι όλες οι προτάσεις θεωρούν ως δεδομένο το Δουβλίνο. Επιμένουν δηλαδή ότι η χώρα στην οποία φτάνει κάποια πρώτο πρόσφυγας είναι η χώρα η οποία ε, θα πρέπει να δεχτεί ή να μην δεχτεί την αίτηση και εντάξει αυτό δεκτό αρκεί να υπάρχει στο σύστημα κάτι το οποίο δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας μηχανισμός αλληλεγγύης ένας μηχανισμός επανεκατάστασης ε, στον οποίο θα συμφωνήσουν να συμμετάσχουν όλες οι χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν δεν γίνει κάτι τέτοιο, ε, κατά με δεν θα μπορέσουμε να λύσουμε το πρόβλημα και θα έχουμε χιλιάδες ετούντες άσυλο οι οποίοι θα αντιμετωπίζονται με τρόπο που κανένας ε, στις χώρες μας ε, δεν θα ήθελε να αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους. Εμείς λοιπόν ως Κοινοβούλιο μπορούμε, όπως κάναμε και στο παρελθόν, να αναλάβουμε την πρωτοβουλία και να ε, ζητήσουμε την εφαρμογή αυτού του μηχανισμού αλληλεγγύης για άλλη μια φορά. Ευχαριστώ. Ωραία. Όταν ξεκινήσαμε τη συζήτηση για το σημείο αυτό, ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου δεν ήταν εδώ. Τώρα είναι εδώ. Να του δώσω το λόγο λοιπόν και να του ζητήσω να μας πει ε, πού βρισκόμαστε με το θέμα αυτό όσο το δυνατόν πιο σαφώς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε που μας ακούτε. Δεν είχα την πρόθεση να μιλήσω σήμερα ε, για αυτό το θέμα, γιατί ε, αύριο ήταν προγραμματισμένο να σας ενημερώσουμε ε, για τις εξελίξεις στο Συμβούλιο και είναι σημαντικό να έχετε μια συνολική εικόνα. Αν ζητάτε σήμερα να σας μιλήσω ειδικά για αυτό το θέμα, να το κάνω. Καταρχάς θα ήθελα να πω ότι εκτιμώ την εργασία της κυρίας Κιγιόμ και τη συζήτηση που έγινε εδώ πάρα πολύ χρήσιμη και δείχνει ότι ε, πράγματι είναι πάρα πολύ περίπλοκο αυτό το θέμα, το θεωρεί και το Συμβούλιο περίπλοκο. Ε, έχει γίνει πολύ έργο στην Ισπανική Προεδρία σε τεχνικό επίπεδο και έδειξε ότι πραγματικά υπάρχουν κάποια θέματα πολύ περίπλοκα και τα αναφέρει και το έγγραφο εργασίας κυρίας Γκυγιόμ αυτά ως Βελγική Προεδρία του Συμβουλίου εμείς συνεχίζουμε τις τεχνικές ε, επαφές στις ομάδες εργασίας του Συμβουλίου και στις αρχές του μηνός διοργανώσαμε μια διπουργική διάσκεψη για το άσυλο και συμμετείχαν και μέλη της Επιτροπής σας για να υπάρχει μια προσέγγιση από τα κάτω προς τα πάνω, από την πρακτική, από την κατάσταση στα κράτη-μέλη προς τα πάνω, αλλά και από οργανισμούς που, που... δραστηριοποιούνται στην κοινωνία για να δούμε ποιες είναι οι διάφορες προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τι περιλαμβάνουν. Όλα αυτά είναι πολύ χρήσιμα και ωφέλιμα για τη δουλειά και του Συμβουλίου, αλλά και τη δική σας εδώ στο Κοινοβούλιο. Λοιπόν, είμαστε διατεθειμένοι να συνεχίσουμε το έργο αυτό στο Συμβούλιο και προσβλέπουμε και στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όπως σας είπα αυτή τη στιγμή και δεν είναι μυστικό άλλωστε, οι συζητήσεις είναι περίπλοκες. Τα πράγματα είναι πολιτικά ευαίσθητα για τα κράτη-μέλη και δεν μπορώ να δώσω αυτή τη στιγμή θέση του Συμβουλίου. Ε, καταλαβαίνετε ότι χρειάζεται συνέχεια στο έργο αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Commissione, la signora Muriel Εξ ονόματο τη Επιτροπή τώρα. Ε, ονομάζομαι Μυριαλ θα ήθελα απλώ να υπογραμμίσω τι παρατηρήσει ε, τη Κομισιόν, να συγχαρώ την κυρία Σιλβί Γκυγιόμ, που όντω και εκείνη υπογράμμισε τα θέματα κλειδιά που αποτελούν αντικείμενο δύσκολων συζητήσεων στο πλαίσιο του Συμβουλίου και που εντόπισε την κεντρική ιδέα των προτάσεων της Κομισιόν που είναι το front-loading, η ενίσχυση της ποιότητας ε, των ε, διαδικασιών σε πρώτου βαθμού για να μπορούν να λαμβάνονται έγκυρες αποφάσεις και θα επιδέχονται λιγότερων επικρίσεων. Ε, να πω ότι αυτή η πρόταση δεν έχει γίνει μόνο για να γίνει ένα ποιοτικό άλμα μέσω νέων διατάξεων, αλλά και επίσης και κυρίως για να αποσαφινιστούν οι κανόνες πρώτης γενεάς, όπου είχαμε διαπιστώσει ότι υπήρχε ανάγκη για περισσότερες ε, κατευθύνσεις και καθοδήγηση. Και για να απαντήσω και στην κυρία Λότφορντ, είναι σημαντικό να θυμίσουμε κάτι, αυτό το σημείο, γιατί έτσι μπορούμε να θέσουμε καλύτερα σε εφαρμογή ένα σύστημα ασύλου πιο αποτελεσματικό. Η κυρία Γκυγιόμ θύμισε το μελλοντικό χρονοδιάγραμμα. Νομίζω πως η συζήτηση έδειξε ότι για να αποφύγουμε αυτό το, το θέμα να ξεχαστεί. Θα πρέπει το Κοινοβούλιο να εκφραστεί γρήγορα, όπως υπενθυμίσαμε και στην Υπουργική Διάσκεψη πριν από λίγες μέρες στις Βρυξέλλες, θα αποτελέσει θέμα κλειδί για τη συνέχιση των, των συζητήσεων. Το ψήφισμα του Κοινοβουλίου για το θέμα αυτό. Μάλιστα. Το λόγο έχει λοιπόν και πάλι η συγχύτρια, η κυρία Γκυγιό. Ναι, κάποιες παρατηρήσεις αγαπητοί συνάδελφοι. Καταρχήν για να απαντήσω στον εκπροσώπους των ε, Ολλανδών ψηφοφόρων της ομάδας της Ελευθερίας, του κόμματος της Ελευθερίας, συγγνώμη, που δεν είχαν έρθει μας στις συνεδριάσεις μας. Όντως θα έπρεπε να έρχονται τα πιο συχνά. Ε, πάντως ε, βλέπουμε πόσο ενδιαφέρον είναι αυτό το θέμα, πόσο σημαντικό είναι απαραίτητα όλα αυτά τα βήματα για τον καθορισμό της ε, δουλειάς που θα κάνουμε για τις άλλες σχετικές οδηγίες. Και ήθελα ακόμη μια φορά να το υπογραμμίσω αυτό. Επίσης, οι περισσότεροι συνάδελφοι μίλησαν για ρεαλισμό και φυσικά και το έχουμε προσέξει. Αυτό μας υποχρεώνει να προσέξουμε περισσότερο και να εστιάσουμε την προσοχή μας στην οδηγία για την ε, διαδικασία. Δεν μπορούμε δηλαδή να μην είμαστε ακριβείς εδώ. Έχω καταγράψει τα όσα ικανοποιούν και τα όσα δυσαρεστούν τους συναδέλφους. Να σας πω μόνο πως γνωρίζω πάρα πολύ καλά, ακόμα και αν σήμερα ακροθυγώς το αναφέραμε, ότι υπάρχουν δυσκολίες για το, θέμα, για το κείμενο αυτό στο Συμβούλιο και γνωρίζω επίσης πως οι συζητήσεις που θα ακολουθήσουν ανάμεσα στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα είναι αρκετά δύσκολες. Υπάρχει πρόβλημα και για το θέμα του κόστους, γιατί το δημοσιονομικό κόστος μια τέτοια συναρμονισμένη ή κοινή πολιτικής που για ορισμένους εκπροσώπους των κρατών μελών είναι ε, δυσθεώρητο. Θα έχουμε την ευκαιρία να επανέλθουμε για όλα αυτά και να δουλέψουμε για το θέμα του κόστους. Αλλά σε αυτό το στάδιο θα ήθελα να σας πω πως είμαι επιπισμένη πως η κακώς ε, χρησιμοποιούμενες διαδικασίες είναι αυτές που κοστίζουν πολύ και κοστίζουν πολύ πέρα από τις διαδικασίες πρώτου βαθμού και όχι τόσο η αύξηση και η εναρμόνιση των κανόνων. Θα μπορούσαμε βεβαίως να, δουλεύουμε, να συνεχίσουμε να δουλεύουμε πάνω σε αυτό το θέμα. ωστόσο, συμμερίζομαι το αίσθημα που εξέφρασαν κάποιοι συνάδελφοι, νομίζω όλοι, το ανέφεραν αυτό, ότι δηλαδή πρέπει να δουλέψουμε με έναν καλό ρυθμό για την υποβολή μιας έκθεσης. Ελπίζω να μπορέσω να το κάνω όσο γίνεται πιο σύντομα παρά τη δυσκολία του θέματος γιατί είμαι επιπισμένη πως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχει μια πολύ ισχυρή θέση για την οδηγία αυτή και για την τροποποίησή της. Δεν υπάρχουν άλλες παρεμβάσεις. Νομίζω ότι είχαμε μια ευρύτατη συζήτηση για ένα ιδιαίτερα δύσκολο και περίπλοκο ζήτημα. Ας ελπίσουμε ότι θα μπορέσουμε σύντομα να καθορίσουμε το χρονοδιάγραμμα για να διασφαλίσουμε ότι θα προχωρήσουν όλες οι εργασίες και θα επιτύχουμε το στόχο μας. Να περάσουμε τώρα στο επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη Σημείο υπαριθμών 6. Γενική προσέγγιση για τις διαβάσεις δεδομένων από τις καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών σε τρίτες χώρες. PNR. Στις 21 Σεπτεμβρίου υιοθετήθηκε ανακοίνωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ε, Γενική Προσέγγιση για τη Διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων, απαντώντας έτσι στο πρόσφατο ψήφισμα του Κοινοβουλίου, το οποίο υιοθετήθηκε το Μάιο. Θα ήθελα να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας παρουσιάσει την ανακοίνωση ε, αλλά να σας υπενθυμίσω τη συζήτηση κυρίως για τα εμπιστευτικά θέματα που αφορούν στις διαπραγματεύσεις στη συμφωνία με την Αυστραλία, τον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες θα γίνει όπως γίνεται συνήθως και κλεισμένο των θυρών. Να δώσω το λόγο λοιπόν στον εκπρόσωπο της Επιτροπής, τον κύριο Πρίμερ, για, τις πρώτες, για την πρώτη παρουσίαση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Όπως είπατε, η Επιτροπή την περασμένη εβδομάδα υιοθέτησε ένα πακέτο προτάσεων για την διαβίβαση στοιχείων των επιθεβατών. Το πακέτο περιλαμβάνει καταρχάς μία